Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αρχίζει και πάλι η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδριάσεως και τα σχετικά κείμενα είναι στη διάθεσή σας. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, ε, γίνονται δεκτά αυτά τα πρακτικά. Ε, έχω να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις ε, σχετικά με τις αντιπροσωπείες ε, ότι στην Επιτροπή Γυναικών δεν θα είναι πλέον μέλος ο κύριος Φιλίπ Ζιμπάν. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις αποδεχόμαστε αυτή την αλλαγή. Το επόμενο θέμα είναι τα θέματα της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και καταρχήν θα συζητήσουμε την περίπτωση του Πακιστάν, τη δολοφονία του Σάμπας Μπάτη, υπουργού των μειονοτήτων και ε, θέλω να δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Λάμπερτς ε, για ε, πρώτη ομιλήτρια ως συντάκτρια του ψηφίσματος. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι μας ήμασταν, ευχαριστήκαμε πάρα πολύ από τη δολοφονία του Υπουργού Σαμπασβάτη είναι γνωστός μας εδώ στο Κοινοβούλιο, έχει επισκεφθεί το Κοινοβούλιο, έχει συναντηθεί με πολλούς από εμά, αλλά επίση επειδή πρόκειται για ακόμα μια συμβολική δολοφονία που χτύπησε κάποιον που αναζητούσε τη συμφιλίωση και δούλευε με όλες τις μειονότητε στο Πακιστάν. Επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε τα συλληπιτήριά μας όχι μόνο προς την οικογένειά του, αλλά προς όλες τις οικογένειες των όσων έχουν δολοφονηθεί σε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Πακιστάν. Μόλις αυτή την εβδομάδα είδαμε δύο τέτοιες επιθέσεις που σκότωσαν πολύ κόσμο. Ο πληθυσμός υποφέρει από εκφοβισμό ε, και υποβαθμίζεται η δημοκρατία στο Πακιστάν. Έχει αλλάξει μάλιστα η δημογραφική κατάσταση σε ορισμένες περιφέρειες, όπως για παράδειγμα στο Κάτα, ε, γιατί ο εκφοβισμός λειτουργεί και διώχνει τον κόσμο. Το ψήφισμά μας ε, θέλει να στηρίξει την ε, δουλειά που γίνεται για την ανοχή και την αμοιβαία κατανόηση και θα έπρεπε να πω ότι το χρειαζόμαστε αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κάποιες υπουργικές δηλώσεις κατά την άποψή μου δεν το βοηθούν αυτό. Αναμένουμε λοιπόν ε, να, πρέπει να παίξουμε λοιπόν ηγετικό ρόλο και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα αυτό και στο Πακιστάν. Ευχαριστώ την κυρία Λάμπερτς, την κυρία Σάκη, τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρόλη την ε, αίτηση του Πακιστανού Υπουργού για προστασία δολοφονήθηκε και αυτό είναι μεγάλη ελοπλήγμα για το Πακιστάν αλλά και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί οι αρχές του Πακιστάν δεν διέθεσαν ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο ή στον Υπουργό ζητώντας ε, να υπάρξει αναθεώρηση εις ε, του νομοθεσία σχετικά με τη βλασφημία προάσπιζε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, ακολουθούσε το παράδειγμα του Υπουργού που είχε δολοφονηθεί επίσης την 1η Μαρτίου. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η ατιμορρησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση και να προσπαθήσει να εφαρμόσει τα μέσα προς ε, επίτευξη δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ την κυρία Σάκ, η κυρία γκεριγγεν Ντεόντεμπερκ ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τον Μάιο του 2010 συζητήσαμε το ζήτημα αυτό στο Στρασβούργο ε, μαζί με τον ε, Υπουργό Σαμπασμπάτη. Το σήμερα μιλάμε για την δολοφονία του. Ε, επίσης, στις 2 Μαρτίου δολοφονήθηκε ένας αξιωματούχος στην χώρα και αυτό μας δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από, την, από τους φανατικούς Ισλαμιστές. Ο Υπουργό δολοφονήθηκε επειδή αγωνιζόταν υπέρ των ε, μειωτήτων και κατά του νόμου περί βλασφημίας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυστυχώς δεν έχει αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Χρειάζεται λοιπόν να οργανώσουμε μια στρογγυλή τράπεζα για το Πακιστάν και για τις μειονότητες. Θεωρώ ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει άμεσα να δράσει και να εξετάσει αυτά τα οποία συνέβη στο Πακιστάν πρωτού χρηνήσουμε νέα θύματα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κόρολα για ένα λεπτό. Ε, η ζωή του κυρίου Μπάτη ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι απειλεί το, το γνώριζε και ο ίδιος ε, και τελικά δεν κατόρθωσε να ξεφύγει. Το Παξανική Βουλή ενέκρινε μια παράξενη τροπολογία του νόμου περί βλασφημίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα σχέσεων ανάμεσα στις ε, διάφορες μειονότητες ε, του Πακιστάν και η ε, τρομοκρατία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία είναι αδύνατον να προστατευτούν υπό το ισχύον κλίμα που επικρατεί στο Πακιστάν. Και ενδέχεται αυτή η κατάσταση να επεκταθεί και σε άλλες γειτονικές χώρες. Ο κύριος Μπάτη ήταν ιδιαίτερα ευφυές άτομο, γνώριζε πολύ καλά τον κινδύνους που διέτρεχε, αλλά χρειάζεται η νομοθεσία του Πακιστάν να τροποποιηθεί και να καταστήσει τέτοιου είδους πράξεις ε, αδύνατες. Ευχαριστώ κύριε Βαντάνε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Πακιστάν πολύ φοβούμε ότι επιδεινώνεται. Υπάρχουν συνεχώς επιθέσεις. Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει καμία επιθυμία να κινηθεί στην αρχή ο, ο στρατηγός Κασίρ είχε ε, δολοφονηθεί και τώρα ο μοναδικός χριστιανός υπουργός Μπάτι δολοφονήθηκε. Συνεργαζόμαστε με το Πακιστάν, ιδίω στο θέμα του Αφγανιστάν. Προσφέρουμε εκατομμύρια ε, ευρώ βοήθεια στο Πακιστάν για να ενθαρρύνουν και τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών. Οπότε θα έπρεπε να ε, είμαστε πιο στεναροί και να πούμε ότι πρέπει να πάψει να υπάρχει προσιλτισμός προς την βία και το μίσος ε, διότι μετά τις πλημμύρες ε, κυβέρνηση της, του Πακιστάν δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημά της και ε, τώρα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Τώρα ο κύριος Σταβάρες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα επίγοντα ψηφίσματά μας πολλές φορές αυτό που μπορούμε εδώ να καταφέρουμε στο Ευρωκοινοβούλιο είναι σχετικά περιορισμένο αλλά τουλάχιστον δύο πράγματα όσον αφορά την ελευθερία έκφραση και την ανεξιθρησκεία σε μια χώρα όπως, το Πακιστάν. Τουλάχιστον δύο πράγματα πρέπει να πετύχουμε στην, ε, στα ψηφίσματά μας. Καταρχήν να πούμε στους υπερασπιστές της ανοχής και της ανεξιθρησκείας στο Πακιστάν ότι δεν είναι μόνοι τους. Αυτό είναι ένας πολύ ταπεινόφρον στόχος, μετριοπαθή στόχος, αλλά τουλάχιστον έχει κάποια χρησιμότητα στη συζήτηση να περάσουμε αυτό το μήνυμα για όσους ε, στο Πακιστάν υπερασπίζουν την ε, ελευθερία πίστης. Και το δεύτερο είναι να πούμε ξεκάθαρα στην κυβέρνηση του Πακιστάν ότι δεν μπορέσει να αφήσει οι φανατικοί στο Πακιστάν να πιστεύουν ότι μιλάνε εξ ονόματο όλων. Γιατί το θέμα της βλασφημίας, όπως αυτό τώρα στο Πακιστάν η κατάσταση που υπήρξε στην Ινδονησία, είναι τόσο παράξενη που πολύ συχνά ε, βαρύνει ολόκληρη μια χώρα επειδή μια μειονότητα φανατικών αρχίζει να μιλά πολύ κραυγαλαία και καταφέρει να επηρεάσει σε του υπόλοιπου. Αν λοιπόν οι κυβερνήσει δεν είναι στην πρώτη γραμμή τη υπεράσπιση τη ελευθερία μέσα στην ίδια του τη χώρα και δεν καταπολεμούν την ατιμορρησία, αν αυτέ ε, οι κυβερνήσει δεν μπορέσουν να σταματήσουν του φανατικού, τότε ολόκληρη χώρα κινδυνεύει να ε, γίνει μία ανεκτική. Αυτό θα πρέπει λοιπόν το μήνυμα να περάσουμε. Όπω τώρα με τη δολοφονία του Υπουργού Μπάτη, όπως και προηγουμένως με τη δολοφονία του κυβερνήτη. Ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε να μην γίνουν έρευνες όπως έγινε με την δολοφονία της πρώην Πρωθυπουργού Μπεναζίρ Μπούτο. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, η κυβέρνηση του Πακιστάν να εξασφαλίσει ότι οι φανατικοί δεν θα ε, τραβήξουν μαζί τους όλο το κοινό και από πολιτική μας πλευρά να στηρίξουμε τους υπερασπιστές της ανοχής στην χώρα αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Ταβάρες. Τώρα έχουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και πρώτα ο κύριος Μάουρο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ο Σέμπατς Βάτη ε, ε, δολοφονήθηκε στο όνομα του υποτιθέμενου νόμου περί βλασφημίας από μια φανατική ομάδα που όπως συχνά συμβαίνει χρησιμοποιεί τον Θεό για να προωθήσει ένα δικό του πρόγραμμα εξουσίας. Ε, με αυτό το ψήφισμα θέλουμε να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Βάτη για την προσπάθειά του όλα αυτά τα χρόνια. Μια τόσο δυνηρή θυσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χρησιμεύσει ως ε, παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε συγκεκριμένες δράσεις να αντικαταστήσουν τα λίγα λόγια που εξάλλου έχουμε εκφράσει με μισή καρδιά μέχρι σήμερα. Μάλιστα τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα το Συμβούλιο και η Επιτροπή αντίθετα από το Κοινοβούλιο έχασαν χρόνο για το αν θα βάλουν ε, τη λέξη χριστιανοί στα καταδικαστικά τους έγγραφα, ενώ οι χριστιανοί εξακολουθούν να σφάζονται βία. Και αυτό γιατί ε, ε, πολύ συχνά μιλάνε για τη Δύση, ενώ για δυτική, δυτικό χαρακτήρα δεν έχει καθόλου αυτή η κατάσταση και γι' αυτό θα πρέπει η Κομισιόν του το να ακολουθήσουν το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Μάιρα. Για ένα λεπτό η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ε, ε, ε, χαιρετήσω την εργασία του κυρίου Μπάτη. Ε, όσοι τον είχαν συναντήσει ε, ε, γνώριζαν πόσο προσπαθούσε να προασπίσει τις μειονότητες στο Πακιστάν και ήξερε ότι η ζωή του κινδύνευε, είχε πολλές απειλές, έχασε τη ζωή του και εμείς χάσαμε εδώ έναν φίλο. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε με το ψήφισμα αυτό. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα ζητούν να υπάρξει ε, σεβασμός της ε, και προστασία της κοινωνίας και ότι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρεται επίσης στο σημείο 19 σχετικά με τα θεσμικά όργανα, την κυβέρνηση του Πακιστάν και τη ρήτρα για τη δημοκρασία και, ε, δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν ε, να συλληπιθούμε και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να στείλει μία προσωπική επιτροπή στο, ε, στη μητέρα του Σάμπας Μπάτη, ο οποίος κυδεύτηκε την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ κυρία Στάιλερ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Γιατεμάκη. Πρόεδρε, η δολοφονία του κυρίου Μπάτη είναι η δεύτερη δολοφονία ενός υψηλά ιστάμενου Πακιστανού μέσα σε δύο μήνες. Ο κύριος Μπάτη και ο κυβέρνητης Τασίτ δολοφονήθηκαν και οι δολοφόνοι του θα πρέπει να ε, βρεθούν, να διωχθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Πέραν από τη δολοφονία του κυρίου Μπάτη θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο καυτό ζήτημα του Πακιστάν η κατάσταση στην ε, επαρχία του Βελουχιστάν Η επαρχία συνεχίζει να υποφέρει από διωγμούς Ξέρουμε πολύ καλά ότι και δεκάδες δικηγόροι έχουν ε, διωχθεί και άλλοι έχουν δολοφονηθεί. Καθώς επίσης ε, δάσκαλοι, καθηγητές, δημοσιογράφοι διώκονται στην ε, επαρχία αυτή. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς το Πακιστάν και να ζητήσουμε από την πακιστανική κυβέρνηση να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Γετεμέκη. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Κιλ Νίλσεν αυτές οι δολοφονίες είναι απαράδεκτες και αυτό που είναι ακόμη πιο απαράδεκτο είναι το συνέστημα τιμωρησίας παρόλο που κλιμακώνονται οι επιθέσεις οι οικογένειες των θυμάτων δεν μπορούν να βοηθηθούν από ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο είναι τελείως διεφθαρμένο βασίζεται δε σε τελείως μεροληπτική εθνικές ε, νομοθεσίες και θα πρέπει να υπάρξει μία μεγαλύτερη εξοπιστία και εντός της χώρας και διεθνώς. Η εργασία την οποία έχει κάνει το Ίδρυμα Heringsberg προσπαθεί να προωθήσει την, την νομοθετική διαδικασία και πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει ό,τι μέτρο έχει για να ενισχύσει τη δικαστική συνεργασία με το Πακιστάν. Ευχαριστώ κυρία Κιλ Νίλσεν. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Τάνοκ. Πρόεδρε, μία μία οι φωνέ μεταρρύθμιση και προόδου εξαλείφονται. Ο Σεμπά Μπάτι γνώριζε ότι, ήταν ότι διέτρεχε κίνδυνο. Εκεί όπου η θρησκευτική δυσανοχή ε, ε, ε, κυριαρχεί σε μια τέτοια χώρα αρνήθηκε να ενδώσει στις απειλές των Ισλαμιστών που τον απειλούσαν ε, με θάνατο. Πριν από ε, λίγους μήνες οι σωματοφύλακες είναι αυτοί που δολοφόνησαν τον ε, κυβερνήτη. Ο Σαμπάτη δεν είχε καν σωματοφύλακες γιατί δεν είχε προστασία ενόπλων ανδρών γύρω του. Αυτή είναι μία από τις ερωτήσεις που θα πρέπει να ρωτήσουμε τον ε, Πρωθυπουργό και είπα τους εκπρόσωπους ελπίζω πως θα θέσει παράδειγμα θα ε, μιλήσει για τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα των εξελίξεων στο Πακιστάν. Ήταν ένας σπουδαίος δημοκράτης. Χαιρετίζουμε τα επιτεύγματα μία ζωή σε αυτή τη συζήτηση και θα πρέπει να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στους δικούς τους αυτή την ε, δυσάρεστη, τόσο δυσάρεστη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο Ισλαμικός νόμος η Σαρία προβλέπει ότι όποιος προσβάλλει το Ισλάμ καταδικάζεται σε θάνατο. Δεν ξέρω εάν ε, αυτή είναι μια σωστή άποψη, πολύ αμφιβάλλω, αλλά οι διάφοροι ακτιβιστές ε, στο Πακιστάν γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το θέμα και το αισθάνονται στο πετσί τους. Ο Σάμπα Μπαχτή, υπουργό της Πακιστανική κυβέρνησης ε, για τις μειονότητε, και ο Μερδίνη ε, κατέστησαν ε, θύματα των εξτρεμιστών στο Πακιστάν. Αυτές οι ομάδες εκφοβίζουν τον λαό αλλά και τους κυβερνήτες οι οποίοι προσπαθούν να μεταρρυθμίσουν το πολιτικό σύστημα. Εν αν ε, δεν ε, επιθυμούμε να επανδρευτούν ε, τέτοια γεγονότα, χρειάζεται να προσπαθήσουμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για έναν επικοδημητικό διάλογο. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία. Μάλλον έχουμε ακόμη έναν εγγεγραμμένο ομιλητή, τον κύριο Ζανέσχη, για ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για την δολοφονία ενός υπουργού, ενός ανθρώπου ο, ο οποίος ε, εκπροσωπούσε τις χριστιανικές του ρίζες, ε, ήταν καθολικός και μιλούμε και για μια δεύτερη δολοφονία στο Πακιστάν που αποδεικνύει ότι οι αρχές αυτής της χώρας δεν ελέγχουν καθόλου την κατάσταση στη χώρα. Αυτή, αυτό είναι πρόβλημα κατά τη γνώμη μου γιατί ουσιαστικά δεν προσπαθούμε να στραφούμε κατά του Προέδρου και της κυβερνήσεως του Πακιστάν. Απλώς λέμε ότι δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ε, την ασφάλεια των ατόμων που έχουν διαφορετική θρησκεία από αυτή που προέχει στη χώρα και κατ' εμέ η κατάσταση στο Πακιστάν χειροτερεύει και πάει. Είναι μια χώρα γεμάτη Ισλαμικό μίσος προς τις ε, άλλες θρησκείες και πρέπει αυτό να καταδικαστεί. Ευχαριστώ κύριε Τζανέσκι. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο και επειδή ορισμένοι πρόεδροι πολιτικών ομάδων και αντιπρόεδροι ε, παρίστανται και συμμετέχουν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι διότι όταν ένα θέμα ενδιαφέρει τόσους πολλούς συναδέλφους θα ακολουθήσω τον ε, κατάλογο και θα σας πω ποιοι είναι οι πρώτοι τους οποίους ε, έχω περιλάβει καταρχάς ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μια εβδομάδα πριν δολοφονηθεί είχα συναντηθεί είχα μιλήσει με τον ε, κύριο Σαμπάς Μπάτη στο γραφείο του στο Ισλαμαμπάκ είχε την εντύπωση ότι δύο στους τελευταίους μήνες και μετά από την δολοφονία του κυβερνήτη του Πουντζάμπ Σαλμάν Τασίρ ε, υπήρχαν πολλές ε, αντιδράσεις και δικηγόροι δημοσιογράφοι δεν τολμούν πλέον να στραφούν κατά αυτών των ε, ε, ε, ακραίων προκλήσεων και παρόλο που είναι συσπηρωμένοι εναντίον της της, ε, ε, της ε, στάσεως αυτής. Αυτός ο οποίος είχε καταργήσει τον νόμο κατά της βλασφημίας είναι ιδιαίτερα σε κίνδυνο και θα έπρεπε τώρα να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος κατά τρόπον ώστε να διακηρύξουμε τη στάση μας εναντίον του εξτρεμισμού. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλε, ο κύριος Άσου για ένα λεπτό. Η δολοφονία του Υπουργού των Μειοτήτων κ. Μπάτη έγινε με βάση τον νόμο περί βλασφημίας. Ο ίδιος ήθελε να τροποποιηθεί ο νόμος. Θεωρώ Λοιπόν, ότι αυτός ήταν και ο βασικός ε, λόγος του δολοφονίας του, αλλά και ο εκφοβισμός τον οποίο υφίστανται όσοι αγωνίζονται για την κατάργηση αυτού του νόμου. Η κυβέρνηση του Πακιστάν χρειάζεται να προλάβει παρόμοιες ε, καταστάσεις ε, στο μέλλον και να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προωθήσει τις δημοκρατικές αρχές που είναι εξάλλου γεγραμμένες στο Σύνταγμά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούτας. Τώρα η κυρία Λεκρύπη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και με τη σειρά μου και εγώ θέλω να εκφράσω την έντονη μου συγκίνηση μετά από την δειλή δολοφονία στις 2 Μαρτίου του Υπουργού του χριστιανού υπουργού κ. Μπατή υπεύθυνου για τις μειονότητες. Αυτή η ομή δολοφονία είναι συνέχεια άλλων δολοφονιών, ε, Πακιστανών, ε, Θαραλέων, ε, υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της γυναίκας. Βλέπουμε λοιπόν ε, θα πρέπει να πετήσουμε από την κυβέρνηση να, ε, να διαφωτίσει αυτή την ε, φρικτή δολοφονία και να εξασφαλίσει αποτελεσματικά την προστασία των ανθρώπων που απειλούνται από τους φανατικούς θρησκευτικούς εξτρεμιστές. Και και σκέφτομαι ε, όχι όλα τα, τις σχετικές ε, οργανώσεις και θα πρέπει με έντονα να ζητήσουμε από όλες ε, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβουν μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση και το Πακιστάν μια ρήτρα σεβασμού της ελευθερίας πίστης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία the Eye, συνάδελφο Τζελίσκα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, τώρα μιλάμε για τη δολοφονία του ε, Υπουργού Σαμπάτη ο οποίος ε, είχε νομοθετήσει το νόμο περί βλασφημίας και ήταν υπέρ της ανοχής η κατάσταση στο Πακιστάν χειροτερεύει συνέχεια και πρέπει να θυμόμαστε τις ε, θρησκευτικές μειονότητες των οποίων τα δικαιώματα καταπατούνται τόσο συχνά. Γι' αυτό και είναι ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να πούμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις διακυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να εφαρμόσουν περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τζιλέσκα ολοκληρώθηκε η διαδικασία Eye και τώρα ερχόμαστε εις ε, την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρουσιάσει ο Επίτροπος και κύριος Χάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον ε, Ιανουάριο είχαμε ε, καταφερθεί ε, κατά της δολοφονίας του κυβερνήτη Σαλμάν Τασίρα αλλά συνέχισε η βία με την δολοφονία στις 2 Μαρτίου του Υπουργού Σαμπάς Μπάτη που ήταν ο Υπουργός υπέρ των μειονοτήτων στο Πακιστάν. Καταδικάζουμε βιαίως ε, την ε, δολοφονία αυτή και ανησυχούμε πολύ για την βία στο Πακιστάν που συνδέεται με τους νόμους περί βλασφημίας. Ο κύριος Αμπάς ήταν πολύ γνωστός, γνωστός για, α, ε, ως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε το θάρρος να καταφέρεται. Παρόλα αυτά ε, τίποτα δεν τον ε, εμπόδισε, ε, δεν του επέτρεψε να υπεραμεινθεί των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό και η κάθε Άστον ζητά από την κυβέρνηση τη Πακιστάν να λάβει τις ευθύνες της και να ε, προστατεύσει όλους αυτούς στην κοινωνία των πολιτών οι οποίοι απειλούνται. Η δήλωση ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να επιβάλλει δικαιοσύνη ε, δεν ε, μας πείθει ότι θα πρέπει συγχρόνως να συλληφθούν ε, και οι υποκινητές και οι εκτελεστές αυτών ε, των ε, εγκλημάτων και στο κλίμα το οποίο υπάρχει μετά την δολοφονία του Σαλμάν Τασίρ βλέπουμε ότι ο νόμος περί βλασφημίας με θανατική ποινή δεν συνάδουν με το πνεύμα που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μας με το Πακιστάν και δεν ενθαρρύνει την δικαιοσύνη και ε, την προάσπιση των μειονοτήτων. Θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε ε, τέτοιες ε, πράξεις τρομοκρατίας άνευ προηγουμένου. Η ελευθερία της θρησκείας είναι ανθρώπινο δικαίωμα, η ελευθερία